της Επιτροπής των Προπολογισμών. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Σας ευχαριστώ όλους ε, για τις ερωτήσεις σας. Οι απαντήσεις ε, διαφώτισαν και το Κοινοβούλιο μας και τις Επιτροπές. Ευχαριστούμε κυρία ε, προτινόμενη Αντιπρόεδρε. Σιγά είχαμε την εντύπωση ότι δεν σας έφτανε ο χρόνος για να μας πείτε ε, τα μηνύματα που είχατε. Λοιπόν, έχετε τώρα στη διάθεσή σας πέντε λεπτά για να συμπληρώσετε τις απαντήσεις σας. Κύριε Αντιπρόεδρε και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τη σαφήνεια των απαντήσεών σας και για τις ε, καταληκτικές σας δηλώσεις. Merci. Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν πω στα καταλεκτικά σχόλια. Με την άδεια των Προέδρων θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Δερμηνείς, όπως πάντα. Είναι καταπληκτική η δουλειά που κάνουν. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αντοχή σας. Uh, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να είμαι πάρα πολύ σύντομη, διότι θα ήμουν άδικη εάν έμπαινα τώρα σε πιο βαθιά ανάλυση και απάντηση ορισμένων ερωτήσεων ε, παραμελώντας κάποιες άλλες που δεν θα προλάβαινα. Πραγματικά και ειλικρινά προβλέπω σε αυτή τη συνεργασία την επόμενη πενταετία θα με έχετε παραστάτη και εταίρος σας σε πάρα πολύ συχνή βάση. Θα ήθελα τελειώνοντας να σας δώσω μόνο δύο μηνύματα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτον, ένα ευχαριστήριο μήνυμα. Όχι μόνο γιατί μου δώσατε το χρόνο σας και μπήκατε σε μια συζήτηση που θεωρώ πάρα πολύ επικοδομητική όσο και καθοδηγητική για μένα και προσανατολιστική. Αλλά σήμερα στην ανταλλαγή απόψεων που είχαμε και με πολλούς από εσά και πριν από την ακρόαση, απεκόμισα την αίσθηση ότι αυτό που μας ενώνουν είναι ακριβώς αυτή η ειλικρινής πεποίθηση ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο μου μήνυμα. Αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ως υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος. Και γνωρίζω ότι θα κάνω πολύ καλύτερα τη δουλειά μου αν κρατήσω ανοιχτά τα αυτιά μου, το μυαλό μου και την καρδιά μου. Και να σας ακούω και να φοβράζομαι και εσάς και το Συμβούλιο, τους λαούς μας. Διότι μπορεί καμιά φορά να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και θα συμβεί αυτό ενδεχομένως. Αυτό θα πρέπει να είναι βάση ο αμοιβαίας ε, συνεργασίας, κατανόησης, να ακούμε ένα τον άλλον για να ενισχύσουμε τα όσα κάνουμε. Σίγουρα κανένας από εμά. Και οπωσδήποτε όχι εγώ. Ούτε το Συμβούλιο, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό τη, ούτε καν το Κοινοβούλιο από μόνος του δεν μπορεί να δώσει αυτή την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στους λαούς μας. Μόνο από κοινού μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα οι τρεις πρόεδροι των Επιτροπών θα πούν και αυτοί κάποια καταληκτικά λόγια. Θα ήθελα προηγουμένως όμως να πω ότι οι συντονιστές της κάθε μια από τις επιτροπές θα συνεδριάσουν από κοινού ε, προπολογισμοί, έλεγχος και γιόρι στις 6 το απόγευμα, 6 με 7.30 στην αίθουσα ASP 1G3. Κυρία Υποψήφια Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ και πάλι σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις μας. Πρώτα απ' όλα τις γραπτές σας ερωτήσεις, αλλά και τις σημερινές, τις 44 ερωτήσεις που σας θέσαμε. Όπως εσείς έτσι και εμείς έχουμε ως φιλοδοξία να κάνουμε ό,τι το καλύτερο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και γνωρίζουμε ότι ο προπολογισμό είναι περιορισμένος, 1% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος. Και ακριβώς επειδή είναι περιορισμένος πρέπει να το συμπεριφερθούμε με πολύ καλό τρόπο, ευγενικά. Είμαστε στην αρχή της θητείας μας και ξέρουμε ποιο είναι το βάρος του παρελθόντος. Η κληρονομιά, 222 δισεκατομμύρια, ε, υπόλοιπα προσεκαθάρισε από το 2013 και 23-24 δισεκατομμύρια απλήρωτοι λογαριασμοί στις 31 Δεκεμβρίου του 2013. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να βρούμε γρήγορα μια διαρθρωτική λύση για να πληρωθούν τα υπόλοιπα αυτά και η Ευρώπη να μην δίνει μια εντύπωση αρνητική εξαιτία του συσσωρευμένου χρέους. Οι δεσμεύσει αυτές αναλήφθηκαν. Πλέον πρέπει να περάσουμε στην πράξη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για τα λόγια σας. Γνωρίζουμε ότι για ορισμένα σημεία θα ήταν πρόωρο να περιμένουμε απαντήσεις, αλλά βλέπετε ήμασταν υπόμονοι μαζί σας. Θέλουμε να αρχίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα η αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, διότι είναι μια μετεκλογική αναθεώρηση. Το πλαίσιο τέθηκε πριν τις εκλογές και σήμερα πρέπει να το καταστήσουμε αρκετά ευέλικτο ώστε να ανταποκριθούμε όσο γίνεται καλύτερα στις προσδοκίες όλων των Ευρωπαίων προσδοκίες για ανταγωνιστικότητα βέβαια, προσδοκίες για ανάπτυξη και προσδοκίες για πλήρη απασχόληση και περισσότερη ευημερία. Αυτά είχα να πω λοιπόν εκ μέρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Βέβαια για τα 300 δισεκατομμύρια θα συζητηθούν ε, πολύ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και αν πρέπει το 2015 να υπάρξει μια δημοσιονομική έκφραση, ελπίζουμε ε, να μας ε, δώσετε τα στοιχεία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γκρέσλερ. Ευχαριστώ πολύ. Να πω κι εγώ το εξής. Κυρία Επίτροπε, το είπατε, ε, μπορούμε να ε, καταφέρουμε καλύτερα, we can do better, το σημειώνουμε αυτό, το παίρνουμε τη μετρητής και να είστε βέβαιοι ότι στο πρόσωπό σας βλέπουμε μία εταίρο για α, μεταρρυθμίσεις. Ε, εδώ και δέκα χρόνια ήταν η πρώτη φορά που η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σπάσει κάποια στεγανά. Προσβλέπουμε σε αυτή σας. Ευχαριστώ. Και εξ ονόματος ε, της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, λέει ο Πρόεδρος κύριος Φόβοντα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ε, Έχουμε τώρα αρκετά στοιχεία και απαντήσεις στη διάθεσή μας για να προχωρήσουμε στην ε, αξιολόγηση. Ραντεβού στις 6, αγαπητοί συνάδελφοι συντονιστές, ε, στην 1G3 του κτηρίου Αλτιέρο Σπινέλη. Ευχαριστώ κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Λήξη συνεδρίες.